και αποφασίζεται έτσι η διάταξη των εργασιών όπως ορίστηκε στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξη. Πριν μπούμε στην ουσία, ε, θα ήθελα μια στιγμή την προσοχή σας παρακαλώ. Θα ήθελα να σας παραπέμψω και να σας θυμίσω την τραγική περίπτωση της Μαλάλα Γιωσαφζάη. Είναι ένα κορίτσι από το Πακιστάν, 14 ετών. Καθόταν στο λεωφορείο και την πυροβόλησε στο κεφάλι ένας Ταλιμπάν τι έγκλημα είχε κάνει. Ήθελε να φοιτούν ε, στο σχολείο τα κορίτσια. Και επιτρέψτε μου στο όνομά σας και ε, του συνόλου του Κοινοβουλίου να εκφράσω τη βαθιά μου συντριβή και να καταδικάσω οξύτατα αυτή τη δειλή πράξη. Καλούμε τις πακιστανικές αρχές να φέρουν τους δράστες ε, στη δικαιοσύνη και να προστατεύουν όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια και να τους ε, εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση. Η κοπέλα αυτή η Μαλάλα εκπροσωπεί συμβολικά πάνω από 250 κορίτσια παγκοσμίω που ζουν στη φτώχεια και δεν έχουν ούτε πρόσβαση ούτε καν προοπτική σε θεμελιώδη στοιχειώδη δικαιώματα όπως είναι η εκπαίδευση. Πριν από δύο εβδομάδες και λιγότερο εορτάσαμε στις 11 Οκτωβρίου την πρώτη Διεθνή ημέρα για τα κορίτσια για να δημιουργηθεί μια συνειδητοποίηση, να καταλάβουμε πόσο συχνά παραβιάζονται τα δικαιώματα των νεαρών κοριτσιών στον κόσμο. Είναι ηθικό μας καθήκον να προστατεύουμε αυτά τα κορίτσια και να τους χαρίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίπτωση της Μαλάλα αισθάνομαι και πατέρας ε, γιατί έχω και μια κόρη και ε, με θλίβει βαθύτατα. Ένα 14χρονο κορίτσι. Τι θέλει, ε, να πάει απλό σχολείο και να αγωνίζεται για να μπορούν και τα άλλα κορίτσια να κάνουν το ε, ίδιο. Αυτό είναι αυτονόητο δικαίωμα, να μπορεί κανείς να φυτέψει στο σχολείο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που να πυροβολούν ένα τέτοιο κορίτσι. εύχομαι σε αυτό το θαραλέο κορίτσι, αυτή τη 14χρονη αγωνίστρια για τα δικαιώματα των κοριτσιών, πλήρη αποκατάσταση της υγείας της. Και ελπίζω ε, ο αγώνας της να εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά νέων κοριτσιών σε όλο τον κόσμο να αγωνιστούμε το ίδιο θάρρος για τα δικαιώματά τους. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, όπως γνωρίζετε κυρίες και